Καταρχήν έλαβα από το ΙΕΦΤΗ e το αίτημα να διοριστεί ο κύριος Μπέλντερ ε, ως μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ιαπωνία στη θέση του, του Μάικ Νάτρασα. Ε, σύμφωνα με το κανονισμό 1.6.4 παράγραφο 2 δεν υπάρχει